Okay, colleagues, shall we start? Ε, ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. So my apologies for the late start. I came rushing from... Συγχωρείτε που καθυστέρησα, ήρθα από μια άλλη συνεδρίαση ως συνήθως. Θα να ξεκινήσω προτείνοντας δύο αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Πρώτα απ' όλα τα σημεία 7 και 8 κοινή συζήτηση για τον κώδικα θεωρήσεων αναβάλλονται. Τα σημεία 9 έως 11 θα τα συζητήσουμε 50 λεπτά νωρίτερα από ό,τι ε, γράφε το αρχικό πρόγραμμα, οπότε όσοι πρέπει να έρθουν για αυτά τα σημεία να υλοποιηθούν. Οπότε αν έχετε κάποιες αντιρρήσεις... Ωραία, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σήμερα λοιπόν έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από την Ιρλανδική. Δεν έχετε κάποια αντίρρηση. Έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω για το τι έγινε στις 26 Απριλίου. Θα τα βρείτε αυτά στα έγγραφά σας. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η κυρία Μποντήλ Βαλέρο ορίστηκε, ορίστηκε εισηγήτρια στην συμφωνία, συμφωνία καθεστώτος Frontex με την Αλβανία και εδώ πέρα λέει απαιτείται συνένεση Πρέπει λοιπόν να δώσει σύμφωνη γνώμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγκρίνει η Επιτροπή τις ε, συστάσεις των συντονιστών. Δεν βλέπω κάποια αντίρρηση. Οπότε μετά έχουμε πράξεις ε, κάτω εφαρμογή και κάτω εξοδότηση. Στις 7 Μαΐου η Κομισιόν ενέκρινε μια πράξη κάτω εξοδότηση που συμπληρώνει την οδηγία 849 του 2015 με κάποιες τεχνικές προδιαγραφές για τα κριτήρια διορισμού κεντρικών σημείων επαφής ε, για παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών πληρωμών. Η βασική νομοθεσία είναι η οδηγία για την πρόληψη της χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θα αποσταλεί λοιπόν η πράξη αυτή σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Έχει το Κοινοβούλιο δύο μήνες για να φέρει κάποια αντίρρηση. Και η εσωτερική μας προθεσμία είναι η 28η Μαΐου στις 12 η ώρα. Αν έχετε λοιπόν κάποια αντίρρηση στείλτε σχετικά στην Πρόεδρο και στην Γραμματεία μέχρι τις 28 Μαΐου, όπως είπαμε. Να τα έχουμε τρεις εφαρμοστικές αποφάσεις ε, της ε, Κομισιόν που επίσης λάβαμε. Η πρώτη περιγράφει μέτρα για την πρόσβαση των δεδομένων στο σύστημα εισόδου-εξόδου και το παράρτημα και το άλλο αφορά την ε, διαγραφή και πρόορη διαγραφή τέτοιων δεδομένων και το τρίτο αφορά την είσοδο τέτοιων ε, δεδομένων ε, στο σύστημα και τα παραρτήματα του. Όλα αυτά είναι ο κανονισμός 226 με συγχωρείτε του 2013. Θα σας ενημερώσουμε και πάλι μέσω του ενημερωτικού δελτίου και πάλι αν έχετε κάποια αντίρρηση ενημερώστε την ε, γραμματεία πριν από τις 21 Μαΐου. Έρχομαστε λοιπόν στο σημείο 3. Έρναμε στην ουσία της ημερήσιας διάταξης. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης ε, της κυρίας ε, Μπαλεστέρο, πρόεδρο του Συμβουλευτικού Φόρουμ της Φροντίκης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και τον κύριο Στέφαν Κέσλερ, πρόεδρο του Συμβουλευτικού Φόρουμ του Frontex για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ανώτερο υπεύθυνο Διαμόρφωση Πολιτική τη Γερμανική Υπηρεσία Ισουητών για του πρόσφυγε. Βεβαίω σα έχουμε ξαναδεί στην Επιτροπή μα. Θα σα δώσω τον λόγο λοιπόν, θα κάνετε μια εισαγωγή και μετά θα γίνει συζήτηση. Κύριε Μπαλιστέρο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι δεν βρισκόμαστε εδώ για πρώτη φορά. Ε, είμαστε πολύ ευγνώμονες πάντα για την πρόσκληση και ε, προσβλέπουμε στη σημερινή συζήτηση. Οι δραστηριότητες μας το 2017. Θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε ένα συμβουλευτικό όργανο στο Frontex το συμβουλευτικό μας φόρουμ, ε, επανελειμμένα τονίζουμε στις εκθέσεις μας ότι δεν έχουμε ούτε την εξουσία, ούτε την εντολή, ούτε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε ε, ή να βεβαιωθούμε ότι ε, εφαρμόζει η Frontex με τέτοιο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα σέβεται όπως πρέπει. Τι κάνουμε όμως, ε, εντοπίζουμε κινδύνους και ενθαρρύνουμε το Frontex να χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία έτσι ώστε να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα ενισχύει στις δράσεις του. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο κάποιες δραστηριότητες και να αλλάζει και η εντολή του Frontex ε, και τώρα προχωράει και η ε, στρατηγική για ένα ενιαίο ολοκληρωμένο έλεγχο και φύλαξη των συνόρων. Τούτων όλων λοιπόν ε, λεχθέντων, επειδή δεν έχουμε και ε, απεριόριστη εντολή, είναι περιορισμένη η εντολή μας, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το ρόλο που διαδραματίζει και η αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Frontex και οι συνεργάτες της για να παρακολουθεί στενά το έργο του Frontex και αυτό είναι πραγματικά κάτι το ε, ευπρόσδεκτο. Έχετε δει όλη την έκθεσή μας που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε σε λίγα λεπτά εισαγωγικά. Θα τονίσω μερικά σημεία μόνο ε, που μπορεί να έχουν κάποιο ενδιαφέρον από την έκθεση πρώτον. Οι επιστροφές. Αυτό συνδέεται με την επέκταση που έχει δοθεί στην εντολή του Frontex και τις δραστηριότητες. 47% δεν απατώμε. Είναι η αύξηση του αριθμού των επιστροφών ε, που έχουν πραγματοποιηθεί. Ως φορούμε έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε παρατηρήσει τρία είδη επιστροφών. Για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επιτόπου παρουσία για να καταλαβαίνουμε πώς εργάζεται ο οργανισμός και να κάνουμε συστάσεις που θα πιάσουν τόπο και θα εφαρμοστούν. Τι παρατηρήσαμε λοιπόν. Είδαμε πώς γίνονται οι επιστροφές. Έχουμε κάνει συζητήσεις και με την διοίκηση του Frontex και τις διαδικασίες για τη φύλαξη των σύνορων για την αρχή της μη ε, επαναπροώθησης στις επανειστοχές και τις επιστροφές. Καταλαβαίνετε ότι λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας του Frontex ε, και το 2019 θα εστιάσουμε σε αυτή την ε, πτυχή. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η στοχευμένη δράση. Όπως αναφέρουμε στην έκθεση, έχουμε συστάσεις για την προστασία των ανηλίκων και ε, αντίστοιχα μέτρα που θα πρέπει να ε, λάβει ε, ο Frontex. Και συνεργαζόμαστε και με την αρμόδια ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ξέρω ότι ήρθε πολύ πρόσφατα στην Επιτροπή σας, η αρμόδια του Frontex είναι μια γενική στρατηγική και γενική πολιτική που θα πρέπει να βοηθήσει το Frontex να καταλάβει ότι η προστασία των ανηλίκων είναι κάτι που αφορά όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της και όχι μόνο ad hoc επεμβάσεις. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει σε όλες τις εργασίες και τη δράση τους. Και το έχουμε ε, επίσης ε, υποβάλει ως σύσταση. Ένα άλλο στοιχείο, το τρίτο, είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ και εσάς ε, που είναι ε, ο μηχανισμός ε, κατάθεσης καταγγελιών ατομικών, προσωπικών καταγγελιών που εγκρίθηκε με το νέο κανονισμό. Εξακολουθούμε να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε το Frontex στην έγκριση ενός νέου εσωτερικού κανονισμού, έτσι ώστε να ενσωματώσει καλύτερα και τις δικές μας συστάσεις και να είναι και ο μηχανισμός αυτός και προσβάσιμος αλλά και να αποδίδει και η αρμόδια του Frontex, όταν ήρθε εδώ στις Επιτροπή σας, αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει εκφράσει ανησυχίες ότι κατατέθηκαν μόνο 19 καταγγελίες, από τις οποίες 5 μόνο θεωρήθηκαν παραδεκτές. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν είναι ε, αντανάκλαση της πραγματικότητας ε, στους ε, τόπους που δραστηριοποιείται η Frontex. Θα το συζητήσουμε αυτό και τη στρατηγική δια διάδοση στην 16η συνεδρίασή μας την άλλη εβδομάδα. Και ένας τέταρτος τομέας πριν δώσω το λόγο στον Στέφαν είναι το ζήτημα του φίλου. Έχουμε εργαστεί στο φόρουμ από το 2015 αλλά και φέτος εκδώσαμε μια σύσταση ε, για την ασωμάτωση ε, του στοιχείου του φύλου ε, σε όλες τις δράσεις του Frontex και προτείνουμε για 10 συγκεκριμένες δραστηριότητες κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν και για ποιο το λόγο το λέω αυτό διότι οι συστάσεις μας βοηθούν το Frontex, είναι καλοδεχούμενες, τους δίνουν συνέχεια και συζητούμε με τη διοίκηση του οργανισμού για το πώς θα υλοποιηθούν ε, το επόμενο διάστημα. Και το εκτιμούμε πολύ αυτό. Υποστηρίζουν πάρα πολύ και τις προτάσεις που κάναμε για το φύλλο και η Frontex στο σύνολο και ιδιαίτερα η αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριος Κέσλερ τώρα. Uh, Uh, Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω την παρουσίαση της έκθεσης αυτής, να παρουσιάσω το δεύτερο τμήμα της ετήσιας έκθεσης για το 2017. Η Μάρτα το ανέφερε ήδη. Όσον αφορά το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, προσπαθούμε εμείς να βοηθήσουμε την αρμόδια θεμελιωδικαιωμάτων να καταφέρουμε να προωθήσουμε όλο και περισσότερο την τήρηση των ανθρωπίνων θεμελιών δικαιωμάτων στα πλαίσια των επιχειρήσεων του Frontex. Ως προς αυτό θα ήθελα να επαναλάβω ένα δόγμα το οποίο έχουμε το οποίο το επαναλαμβάνουμε μάλιστα συνεχώς και ενώπιον τη δική σας επιτροπής. Ζητούμε να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα, το απαραίτητο προσωπικό και απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει σωστά το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Frontex. Αυτή τη στιγμή, κάτω από το 2% του οργανισμού απασχολείται για το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεδομένη αυτή τη στιγμή τη διευρυμένης εντολής και των περισσότερων αποστολών που προβλέπονται για το Frontex, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καταφέρουμε να έχουμε το απαραίτητο προσωπικό και την απαραίτητη χρηματοδότηση. Ιδίω αν δούμε επίση και τι ε, σημαντικότερε πλέον επιπτώσει που έχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα οι δραστηριότητε και επιχειρήσει του Frontex. Θα ήθελα επίση να τονίσω ότι το μεγαλύτερο μέρο του προσωπικού που εργάζεται στο Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι άνθρωποι που παρέχουν κυρίω τεχνική υποστήριξη. Το Γραφείο Θεμελιών Δικαιωμάτων απασχολεί προφανώ και κάποιου εργαζόμενου οι οποίοι ασχολούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτά καθεαυτά, αλλά πιστεύουμε ότι ο αριθμό των εργαζομένων αυτών θα πρέπει να ενισχυθεί, θα πρέπει να αυξηθεί. Νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περισσότερου πόρου, χρηματικού και ανθρώπινου, προκειμένου να καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρας πιο αποτελεσματικά το έργο μας. Αυτό είναι αίτημα το οποίο το έχουμε επαναλάβει και στο παρελθόν και το υποβάλλουμε εκ νέου. Δεύτερον, Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει ο Frontex να συνεργαστεί περισσότερο με τρίτες χώρες. Έχουμε την Τουρκία και τη Λιβύη που αποτελούν ε, εξαιρετικά παραδείγματα τη συνεργασία που θα μπορούσαμε να έχουμε στο μέλλον για την περαιτέρω προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στι επιχειρήσει του Frontex. Το αναφέρω απλώ αυτό αυτή τη στιγμή και ενδεχομένω να βαθύνουμε περισσότερο κατά τη διάρκεια τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Στα πλαίσια των επιχειρήσεων του Frontex αυτό που μας ε, ενδιαφέρει περισσότερο κατά το 17 ήταν να επιμείνουμε περισσότερο στην περιοχή της Μεσογείου και να εγκρίνουμε ένα κώδικα διοντολογίας για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εμπλέκονται σε δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης. Ως προς αυτό, τονίζω για μία ακόμη φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οποιοδήποτε φορέα εμπλέκεται σε τέτοιε δραστηριότητε έρευνα και διάσωση, θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την προστασία των μεταναστών, των προσφύγων που επιβαίνουν σε σκάφη. Αυτό αποτελεί, θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Παράλληλα, το φόρουμ έχει τονίσει περισσότερο το ζήτημα των θεμελιών δικαιωμάτων σε σχέση με τις επιχειρήσεις της Frontex στην Ουγγαρία όπου βλέπουμε ότι η πρόσφατη έγκριση μιας νομοθεσίας στη χώρα αυτή έχει θέσει εν κινδύνο τα θεμελιώδη δικαιώματα σε αυτή τη χώρα στα πλαίσια των επιχειρήσεων της Frontex. Επίσης, προβλέπεται και η αναθεώρηση της στρατηγικής θεμελιωδών δικαιωμάτων του Frontex Ξέρετε ότι ε, αναμένεται από το Frontex να καταρτήσει μια στρατηγική, μάλλον είχε καταρτήσει στο παρελθόν μια στρατηγική θεμελιωδών δικαιωμάτων ο Frontex όπως το γνωρίζετε. Καλείται αυτή τη στιγμή να αναθεωρήσει αυτή τη στρατηγική. Περιμένουμε ακόμα να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της αναθεώρησης αυτής. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε κι εμείς να εμπλακούμε στην αναθεώρηση αυτή, προκειμένου να συνεχίσουμε και φέτος και στο μέλλον να προασπιζόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει πραγματικά στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής να αντανακλάται ε, η εντολή και οι ικανότητες ε, του ε, οργανισμού του Frontex, που θα πρέπει πάντα να προβλέπει την καλύτερη δυνατή τήρηση και προάσπιση των θεμελιδών δικαιωμάτων. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι πάρα πολλοί βουλευτές παρόντες σήμερα. Νομίζω όμως ότι όλοι όσοι είναι παρόντες θέλουν να πάρουν το λόγο για το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα θέμα το οποίο είχε να κάνει με τις ε, θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά μας ε, αναστατώνει αυτή τη στιγμή το ότι ε, ακούμε ότι δεν έχετε τα απαραίτητα μέσα. Εφτά θέλουν να πάρουν το λόγο. Σύπελ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την παρουσίαση της έκθεσης. Μετά από τα σχόλιά σας, Έχω καμία φορά την αίσθηση ότι το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι ένα για ό,τι άλλο συμβαίνει στη Frontex. Και γιατί το λέω αυτό. Δύο ερωτήσεις, έχω, μάλλον δύο ζητήματα. Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εμφανή απροθυμία του Frontex να ε, στελεχώσει όπως θα έπρεπε το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σήμερα δεν είναι σε θέση οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους εκεί. Και μεταξύ αυτών είναι και η παρακολούθηση ε, κάποιων υποχρεώσεων που έχουν από την εντολή του Frontex για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και το δεύτερο, το και οι δύο μιλητές, υπάρχουν ακόμα περιορισμοί στην πληροφόρηση που έχει το δικό σας φόρουμ, ιδιαίτερα πληροφόρηση ε, σε σχέση με τις επιχειρησιακές ε, δράσεις και τα διάφορα μέτρα. Πρέπει να βρεθούν λοιπόν λύσεις και τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξουμε το έργο σας και να βρούμε μια λύση σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα και Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέστερ. Uh, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Η ετήσια έκθεση του Συμβουλευτικού Φόρουμ λέει ότι η Frontex έχει μειώσει σημαντικά τον αριθμό των ανδρών που έχει αναπτύξει. Υπάρχουν δημόσιες πληροφορίες για τον αριθμό των ατόμων που παραμένουν στην Ουγγαρία. Έχουν ληφθεί ανάλογα μέτρα στην Κροατία, όπου έχουμε τακτικές παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων όπως ε, καταγγέλουν διάφοροι τα τελευταία χρόνια. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex είπε πως η παρουσία της Frontex θα μπορούσε να συνεισφέρει στο να μειωθεί η χρήση βίας στα σύνορα αλλά και στην καταγραφή των γεγονότων επιτόπου. Γνωρίζετε αν η Frontex κατέγραψε περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά ετούντων άσυλο στην Ουγγαρία ή στην Κροατία. Εάν ισχύει αυτό, υπάρχουν κάποιες ε, δημόσιες εκθέσεις. Όπως σωστά είπε το Φόρουμ, οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν επιτείνει τον κίνδυνο η Frontex να εμπλεκεί σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 2017. Πάνω από 3.000 Εκατό μη σύνομες αποθήσεις έγιναν από την Ουγγαρία, προς τη Σερβία. Πάνω από 1.100 άτομα απελάθηκαν από τη χώρα. Σύμφωνα με εκθέσεις της υποθαρμοστίας του επιπλέον, οι ακτιβιστές έχουν καταγράψει πολλές ε, περιπτώσεις ε, αξιωματούχων της ε, Frontex που συμμετείχαν ή ήταν μάρτυρες υπερβολικής βίας γνωρίζει το φόρουμ τέτοια γεγονότα. Υπάρχουν στοιχεία για τέτοιες περιπτώσεις στα εσωτερικά έγγραφα τη Frontex. Ποια είναι η αντίδραση της υπηρεσία σε αυτέ τι ε, κατηγορίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κινίτσι. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο καλεσμένους μας και να τους ευχαριστήσω κυρίως ε, όχι μόνο για λόγους ευγένειας αλλά επί της ουσίας πραγματικά γιατί ε, ασχολήθηκαν στα πλαίσια της έκθεσής τους με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, ζήτημα το οποίο με απασχολεί όλους ιδιαίτερους, ιδίως όσον αφορά τους ανήλικους, τα μικρά παιδιά, τα οποία θα πρέπει πάντα να τα προστατεύουμε. Τονίστηκε μάλιστα στην αρχική παρέμβαση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πλέον μια σφαιρική στρατηγική προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε σφαιρικά τους ανήλικους μετανάστες και πρόσφυγες. Ξέρετε ότι στην επέτειο αυτή της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ψηφίσαμε και ένα ψήφισμα στο, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου όπου ζητάμε εκ νέου να μπορούμε να προστατεύουμε πιο αποτελεσματικά με άμεση εφαρμογή τα δικαιώματα των ανηλίκων. Σε σχέση με αυτό λοιπόν θα ήθελα να κάνω την ακόλουθη ερώτηση. Ποια προβλήματα ακόμα θεωρείτε ότι υπάρχουν όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς προκειμένου να σας βοηθήσουμε εσά με το έργο σας και προκειμένου οι ανήλικοι να χαίρουν τις πλήρους προστασίες που τους αρμόζει. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους προσκεκλημένους μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας ε, δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση που βλέπετε στην Λιβύη. Έχουμε μια κατάσταση για την οποία τα κράτη-μέλη είναι σε άρνηση και όχι μόνο τα κράτη-μέλη. Ε, και τα θεσμικά όργανα παριστάνουν ότι εκπαιδεύουν ε, τις ντόπιες δυνάμεις, ενοπλές δυνάμεις ε, να βοηθήσουν την αντιμετώπιση προσφύγων και μεταναστών, αλλά γνωρίζουμε πως πρόκειται περί κατσαπλιάδων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να καταστήλουν πρόσφυγες και μετανάστες. Αν μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες ε, για να μπορέσουμε να επισημάνουμε τις ευθύνες ε, των κρατών μελών που αρνούνται την πραγματικότητα στην Λιβύη. Γνωρίζετε ε, το τι συμβαίνει. Και στην Ουγγαρία ο κύριος Κέσλερ ανέφερε την κατάσταση στην Ουγγαρία όπου όντως η Frontex ε, όπως είπατε κινδυνεύει να εμπλακεί σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, για τις οποίες είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση της χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα, να μας πείτε περισσότερα για το ποια είναι η δική σας εικόνα. Η κυρία Σπινέλη. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τους δύο καλεσμένους για τις δύο αυτές παρεμβάσεις. Και όπως είπε και η συνάδελφος Σίπελ, έτσι και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας τρόπος για να αποφύγουμε πλέον όλα αυτά τα άλοθη και να αρχίσουμε επιτέλους να μιλάμε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, σαφήνεια και διαφάνεια, ζητώντας περισσότερο προσωπικό και μεγαλύτερη πρόσβαση σε τεκμήριωση, όπως είπατε. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα σημεία τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να θίξουμε που χρειαζόμαστε ουσιαστικά μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια με τη δική σας ε, τη συμβολή όσον αφορά την ε, επαναπροώθηση που γίνεται προς τη Λιβύη. Στην έκθεσή σας αναφέρεστε σε κάποιες ανησυχίες, concerns στα αγγλικά, αλλά δεν ακριβώς και αναφέρεστε εδώ πέρα σε κάποιες οργανώσεις ε, συμπεριλαμβανομένες μιας οργάνωσης που συμμετέχει και στο δικό σας το φόρουμ. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η οργάνωση αυτή που συμμετέχει στο δικό σας το φόρουμ και η οποία εξέφρασε ανησυχίες και ποιες είναι ακριβώς αυτές οι ανησυχίες, γιατί δυστυχώς δεν γίνεται ρητή αναφορά στην εκθεσή σας. Μιλάτε για φαινόμενα βίας, μιλάτε για κατάχρηση, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε και δολοφονίες, φαινόμενα δουλείας, έχουμε βιασμούς. Δεν νομίζω λοιπόν μπορούμε να αρκεστούμε πλέον σε γενικόλογες εκφράσεις, πρέπει να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Ένα άλλο σημείο νομίζω επί του οποίου χρειάζεται μεγαλύτερη πάλι σαφήνεια είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο ότι διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή ότι μειώνονται οι αφήξεις στην Ευρώπη, ενώ από την άλλη βλέπουμε ότι αυξάνονται οι θάνατοι στη θάλασσα. Οι δύο αυτοί παράγοντες ε, αναφέρονται τελώς ξεχωριστά στην έκθεσή σας. Επίσης δεν κάνετε ρητή αναφορά στους θανάτους στη θάλασσα, ενδεχομένως να είναι περισσότερο το 2018. Όντως είχαμε μια ρητή αύξηση, σαφή αύξηση των θανάτων το 2018 στη θάλασσα. Και μία ακόμα ερώτηση όσον αφορά την πρόσφαση σε πληροφορίες σε σχέση πάντα με την ακτοφυλακή, με τις δυνάμεις της ακτοφυλακής. Πριν από δύο εβδομάδες, ένας εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σωματείας Shell είπε εδώ πέρα στην Επιτροπή μας σε σχέση με τον μηχανισμό παρακολούθησης πιθανής καταπάτησης θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επιχείρηση Σοφία. Είπε λοιπόν ότι το Συμβουλευτικό Φόρουμ έλαβε μία έκθεση για τον μηχανισμό παρακολούθησης. την έκθεση αυτή, εσείς την έχετε λάβει, πραγματικά είναι διαθέσιμη για το κοινό. Δεν διευκρινίστηκε αυτό στην παρουσίαση που έγινε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κέλλερ, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το έργο σας. Το διαρκές εκεί στο Συμβουλευτικό Φόρουμ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως το είπατε, και η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο ολόκληρο έχει αγωνιστεί για να υπάρχει υπεύθυνος για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο Frontex. Δεν θα υπήρχε ε, χωρίς το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας. Μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Αν δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της, κύριε αυτή, επειδή δεν είναι καλά στελεχωμένη η υπηρεσία της. Θυμάστε ότι και για να οριστεί η ίδια ε, χρειάστηκε να πιέσει η Επιτροπή μας, για να το πω έτσι φιλικά. Μήπως θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Ε, να τονίσουμε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο θεσμός. Και το δικό σας φόρουμ και η αρμόδια για το θεμελιώδη δικαιώματα. Μήπως ο πρόεδρος της Επιτροπής να στείλει καμία επιστολή στο Frontex λέγοντας ότι οι θέσει θα πρέπει να πληρωθούν, να στελεχωθεί σωστά αυτή η υπηρεσία και το συμβουλευτικό σα φόρουμ να παίρνει όλη την ενημέρωση που χρειάζεται, τα διάφορα έγγραφα που λέτε στην έκθεσή σα, τα οποία δεν έχετε πρόσβαση. Και επίση οι ειδικέ σα συστάσει δεν θα πρέπει να αγνοούνται. Γιατί τι να το κάνω να έχω συμβουλευτικό φόρουμ όταν συμβουλεύει και δεν το λαμβάνει κανεί υπόψη, ή σχεδόν ποτέ ας πούμε στη στρατηγική για το φύλλο είναι πολύ ωραία αυτά που λέτε, αλλά αν δεν εφαρμόζονται είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνετε κάποια συνέχεια, μη τι άλλο να το συζητάνε. Δεν λέω να το υιοθετήσουν 100% προφανώς, συμβουλευτικό όργανο είστε, αλλά τουλάχιστον να το συζητούν. Έτσι ώστε να σέβονται τη δουλειά σας και να μείνουν συνέχεια και να την αντιμετωπίζουν σοβαρά. Άρα θα πρότεινα να γράψει ο πρόεδρος μια επιστολή στο Frontex και να αναφέρει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας ή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο να λειτουργούν σωστά αυτές οι δομές και οι θοσμοί. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να θέσουμε μεγάλες εκθέσει και το Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω, αυτό που είπατε για τη συνεργασία του Frontex με τι τρίτε χώρε και πόσο σημαντικό θα ήταν να έχουμε μια εκτίμηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα πριν ε, από τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών με τρίτες χώρες. Και σε εκθέσεις για το Frontex και τις τρίτες χώρες αυτό θα το λάβουμε υπόψη, οπωσδήποτε θα παίξει ρόλο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Um, κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών επισκέφθηκε τα βουλγαροτουρκικά σύνορα προσφάτως. Είδαμε και τους συνοριοφύλακες και την επιχείρηση της Frontex. Και αυτό το οποίο μας είπε η κοινωνία των πολιτών στη διάρκεια της αποστολής μας είναι ότι όταν η Frontex είναι μέλος ε, του περιπόλου ακολουθούν ε, τα προβλεπόμενα. Όταν δεν είναι στις περιπολίες ε, προκύπτουν προβλήματα. Αναρωτιέμαι. Το θέμα της νομιμοποίησης μιας κατάστασης αποτελεί ποτέ αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ημών και της ηγεσία της Frontex, γιατί αυτό το οποίο κατάλαβα εγώ από την επίσκεψη στη Βουλγαρία είναι ότι επειδή η Frontex δεν κάνει ποτέ ευνηδιαστικούς ε, έλεγχους ή μάλλον ε, περιπολούς και είναι κατόπιν ε, προσκλήσεως των εθνικών αρχών της Βουλγαρίας προκειμένου και βεβαίως δεν έχουν ως στόχο την, τον έλεγχο των διαδικασιών αλλά βρίσκονται εκεί πέρα για να γνωρίζει ο κόσμος ότι ο έλεγχος των συνόρων γίνεται με βάση κάποιες προδιαγραφές, κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν γίνεται. Το άλλο θέμα είναι η κατάσταση με την Ουγγαρία, όπου είπατε ότι ίσως δεν θα έπρεπε η Frontex να συνεχίσει να δραστηριοποιείται εκεί και αντιλαμβάνομαι ότι πράγματι υπάρχει μια περιορισμένη παρουσία της Frontex επί αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί και ασκήσατε κριτική. Δεν έχω καταλάβει τι ρόλο μπορεί να παίζει η Frontex σε εξωτερικά σύνορα Σέγγεν με ένα πολύ μεγάλο φράχτη και πολύ περιορισμένη εισρωή. Γιατί δηλαδή να είναι εκεί ακόμα η Frontex. Μπορείτε να μου εξηγήσετε το σκεπτικό που έχουν ή αυτοί είτε η ε, κυβέρνηση εξωτερικής. Ναι, καταντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε με τη στάση του σώματός σας, αλλά θα επιμείνω στην ερώτηση μου. Ε, έχουμε μετά την τρίτη ερώτηση. Όταν συστάθηκε η συνόρια φυλακή και ακτοφυλακή υπήρχε αυτή η συζήτηση για το Εάν τα κράτη-μέλη δεν φύλαγαν τα σύνορά τους με τρόπο που θα άρεσε σε άλλα και τότε θα υπήρχε η δυνατότητα να αναλάβει δράση από μόνη της η συνοριοφυλακή. Κάτι το θεωρητικό βεβαίως γιατί εξακολουθούσε να είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους. Μπορείτε ίσως να μου εξηγήσετε ποια είναι η σχέση μεταξύ των κρατών μελών και του γραφείου της Frontex στην Βαρσοβία με τον νέο αυτόν τρόπο αντιμετώπιση των ευθύνων. Και τέλος θα ήθελα να επεκταθείτε στις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Άκουσα συναδέλφους να ρωτάνε για την Λιβύη και την Τουρκία. Αλλά ακούσατε μόλις ε, πως έχουμε μία έκθεση για την συμφωνία Frontex Αλβανίας και εδώ πέρα θεωρώ ότι αναθέτουμε σε τρίτη χώρα τους συνοριακούς μας ελέγχους παρουσία ε, μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Ε, τι ρόλο παίζουν εκεί. Σας ευχαριστώ κύριε Γιουρέκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και η ερώτησή μου έγινε ε, ήδη από την Αναγκόμες. Ε, ε, ήθελα δηλαδή να σας ρωτήσω τον κύριο Κέσλερ συγκεκριμένα να αναπτύξει λίγο αυτές τις ιδέες περί παραβιάσεως ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Frontex στα Ουγγρικά σύνορα. Τι δραστηριότητες εννοείται. Και κατηγορίες ε, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι άνδρες της ε, Frontex και οι γυναίκες βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Πριν επανέλθω στους ομιλητές μας, ε, να πω και εγώ δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα αναφέρατε το ότι η Frontex ε, δεν θέλει να επιβάλλει τις ε, συστάσεις ε, περί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Άννα Γκόμες είπε ότι τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε μια κατάσταση άρνησης. Ε, συμβαίνει το αντίθετο, ότι είναι τμήμα, δεν θα πω της στρατηγικής, αλλά της προσέγγισης των κρατών μελών, γιατί η συμφωνία με την Λιβύη ε, δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε κατά λάθο. Ε, έβαλαν την υπογραφή τους ε, τα τη άρα συμφωνούν. Δεν υπάρχει καμία άρνηση δηλαδή. Ε, κάτι το οποίο έγινε και εμένα. Και έρχομαι εδώ στη δεύτερη ερώτηση ή παρατήρηση. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα λύσει το όργανο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι θέμα των πολιτικών, αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις, οπότε βέβαια το βάρος πέφτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμφωνώ εδώ πέρα με την πρόταση της ε, Σκακέλερ. Ο Κλοντ Μωραές δηλαδή να απευθύνει μια επιστολή εξ ονόματος της ε, Επιτροπής μας που θα καλύπτει διάφορα ζητήματα. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν ε, επαρκείς δυνατότητες, ότι δεν υπάρχει στελέχωση, αλλά και γενικότερα να δούμε το πώς εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τι γίνεται με αυτές τις συμφωνίες. Και νομίζω μπορούμε να δούμε και τον προπολογισμό και να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη στήριξη. Λοιπόν, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε. Λοιπόν, πολλές και πολύπλοκες οι ερωτήσεις που θέσατε και δεν είμαι πεπισμένος θα καταφέρουμε να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις επαρκώς. Και αυτό διότι θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι εμείς δεν είμαστε οργανισμός παρακολούθησης και επιτήρησης της Frontex. Δεν επιτηρούμε εμείς τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μολονότι μερικές φορές μου δίδεται η εντύπωση ότι έχουμε εμείς ακόμα λιγότερες πληροφορίες για ορισμένα ζητήματα από ό,τι είχετε εσείς. Θα ήθελα τώρα να επισέλθω σε κάποιες λεπτομέρειες, κύριο Κέστερα. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα όσον αφορά τους αξιωματούχους που έχει η Frontex στην Κροατία και την Ουγγαρία. Νομίζω ότι το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το υποβάλλετε στους ίδιους αξιωματούχους της Frontex. Εμείς δεν έχουμε καθημερινά στατιστικά δεδομένα όσον αφορά τους αποσπασμένους στις χώρες αυτές αξιωματούχους της Frontex στα πλαίσια των επιχειρήσεων του οργανισμού. Επίσης, δεν γνωρίζουμε και το λέω αυτό με απόλυτη συνείδηση. Δεν γνωρίζουμε για κάποια έκθεση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που να έχει συντάξει Frontex ή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που να έχει γίνει από τη Frontex. Δεν μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν υπήρξαν τέτοια περιστατικά. Πάντως, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία επίσημη τεκμηρίωση, καμιά τέτοια επίσημη έκθεση της Frontex για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρατε στα περιστατικά εκείνα που έχουν να κάνουν με την Κροατία. Το σύντημα αυτό μας έχει απασχολήσει και εμάς Θεωρούμε πάντως ότι τα συμβάντα αυτά δεν έγιναν στα πλαίσια των επιχειρήσεων της Frontex. Και ξέρετε ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την εντολή για να διερευνήσουμε περαιτέρω τα περιστατικά αυτά. Για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω ότι είμαστε ένα συμβουλευτικό όργανο στα πλαίσια της Frontex. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εμεί μια σφαιρική εικόνα όλων των πτυχών των επιχειρήσεων της Frontex στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις της κυρίας Γκόμες. Για άλλη μια φορά, σας τονίζω ότι δεν έχουμε εμείς τις δικές μας πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση στη Λιβύη. Προφανώς έχουμε πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μας ενημερώνουν για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λιβύη και νομίζω ότι αναφέρατε εσείς ήδη τις πληροφορίες αυτές που έρχονται από την Human Rights Watch ή την Amnesty International. Δυστυχώς όμως εμείς δεν έχουμε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες από τις δικές μας πηγές, ακριβώς επειδή δεν έχουμε τις πηγές αυτές τις δικές μας επιτόπου. Πάντως νομίζω ότι θίξατε κάτι πολύ σημαντικό. Ζήτημα το οποίο μας είχε απασχολήσει και μας πολύ συχνά στο παρελθόν. Κατά την άποψή μας, ο Frontex θα πρέπει να κάνει μια σφαιρική αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του καθεστώτος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προτού συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες. Και αυτό προφανώς ισχύει και για τις συμφωνίες για το καθεστώς Frontex, όπως αυτή που πρόκειται να συζητήσετε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλβανίας. Δεν νομίζω ότι προβλέπεται, από όσο ξέρω τουλάχιστον, μια αξιολόγηση κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία προτού συναυθεί η συμφωνία αυτή. Επομένως, πάλι δεν μπορώ να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση περαιτέρω πληροφορίες. Κυρία Σπινέλη, τώρα απευθύνομαι σε εσά. Η επιχείρηση Σοφία, στην οποία αναφερθήκατε, με επιχείρηση αυτή δεν αποτελεί επιχείρηση της Frontex. Συνεπώς, για άλλη μια φορά, στα πλαίσια της Frontex τουλάχιστον δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένε πληροφορίες, δεν μπορώ να κάνω καν σχόλια σε σχέση με το τι γίνεται στις επιχειρήσεις Σοφία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο η δική σα Επιτροπή θα μπορούσε να θίξει. Το γεγονό, δηλαδή ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντε, οι οποίοι διεξάγουν πολλέ διαφορετικέ επιχειρήσει, χωρί να υφίσταται κανένα ενιαίο καθεστώ ανταλλαγή πληροφοριών, χωρί να υπάρχει καμία σφαιρική παρακολούθηση, κανένα φορέα ο οποίο θα μπορούσε να δει πραγματικά ποιο είναι ο αντίκτυπο των επιχειρήσεων αυτών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω και πρωτού δώσω το λόγο στη συνάδελφο την Μάρτα. σε σχέση με τα σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Αναφερθήκατε σε ένα επιχείρημα το οποίο ακούμε πολύ συχνά και σε σχέση με άλλες χώρες. Αν ο Frontex είναι παρόν επιτόπου, αν έχει γραφεί επιτόπου σε μια χώρα, τότε σαφώς έχουμε έναν καλύτερο έλεγχο του τι συμβαίνει επιτόπου από το να μην είμαστε εκεί. Το θέμα αυτό το συζητήσαμε και στα πλαίσια της ε, Ουγγαρίας. Εμείς είχαμε πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το να έχει κανείς άμεσα πληροφορίε οι οποίες να προέρχονται επί τόπου, αλλά αν δεν τις αξιοποιούμε τις πληροφορίες αυτές εν συνεχεία, τότε δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε πληροφορίες που έρχονται επί τόπου από την παρουσία που έχει η Frontex επί τόπου, τότε είναι καλύτερο να αποσύρεται η Frontex από μια χώρα από το να παραμένει. Και προσοχή, δεν αναφέρομαι αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένα συμβάντα τα οποία μπορούν να έχουν να κάνουν με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω των γραφείων της Frontex στην Ουγγαρία. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι ε, η παρουσία της Frontex στη χώρα αυτή, η οποία ήταν όντως περιορισμένη, η παρουσία πάντως της Frontex στη χώρα αυτή λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο όπου ε, η τήρηση και προάσπιση των δικαιωμάτων δεν την χάνει πλέον κάποιε εγγύησει. Επομένω αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει εμά είναι να γνωρίζουμε τι κάνει η Frontex προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια των περιστάσεων που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην Ουγγαρία. Δεν έχουμε πάλι συγκεκριμένε πληροφορίε για κάποιο συγκεκριμένο συμβάν. Εμεί αναλύουμε απλώ το γενικό πλαίσιο και λέμε βάσει των πληροφοριών αυτών, βάσει της ανάλυσης που κάνουμε του πλαισίου αυτού, θεωρούμε ότι η Frontex θα ήταν καλύτερο να αποσυρθεί από την να συνεχίσει να παραμένει επιτόπου. Thank ε, Κυρία Παλαιστέρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπε και ο Στέφαν, είμαστε σε πάρα πολύ δεινή θέση. Μας κάνατε πολλές ερωτήσεις, αλλά Ταυτόχρονα βεβαίως ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Διαβάζετε την έκθεσή μας, προβληματίζεστε, κάνετε προτάσεις, ερωτήσεις. Και η ίδια μας η ύπαρξη ε, εξαρτάται πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη σχέση από το Κοινοβούλιο και ορισμένες ε, πρόοδοι ε, στη λειτουργία του Frontex έχουν γίνει μόνο χάρη στη δική σας υποστήριξη και παρέμβαση. Ε, Χαίρομαστε και για τις συγκεκριμένες προτάσεις. Ρωτάτε τι μπορείτε να κάνετε. Για τη στελέχωση του γραφείου θεμελιωδών δικαιωμάτων, τι κάναμε εμείς, ρωτήσαμε την ίδια την επικεφαλής, τι ανάγκες έχετε, ποιες είναι οι ελάχιστες ανάγκες για να μπορείτε να λειτουργείτε σωστά να ανταποκρίνεστε στις ευθύνες που έχετε και στην εντολή. Να δούμε ποιες θέσεις θα είναι αυτές στο οργανόγραμμα ε, και σε τι βαθμό και σε τι επίπεδο είναι αυτή η υπάλληλοι. για να μπορεί να λειτουργεί σωστά η υπηρεσία. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση και στις πληροφορίες, κοιτάξτε τι σημαίνει εδώ. Είναι περίπλοκο αυτό. Βεβαίως. Εμείς πολλές φορές ε, έχουμε πληροφόρηση, υπάρχουν και κάποια έγγραφα, καταλαβαίνετε ότι είναι διαβαθμισμένα και μπορεί να μην έχουν μεγάλη σχέση με τη δική μας δουλειά. Κάνουμε επισκέψεις, αν, ανέφερα, επισκέψεις που κάναμε σε επίπεδο επιστροφών, που είχαμε την ενημέρωση, την απαραίτητη και αυτή που χρειαζόμαστε εγκαίρως λειτουργούν σωστά. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου θα περιμέναμε ε, πιο έγκαιρη ενημέρωση και αυτό δεν συμβαίνει. Όπως και σε άλλε εξελίξεις που απευθυνόμαστε σε εσά για να δούμε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Εμείς από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να το συζητούμε αυτό επικοδομητικά με το Frontex για να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο λειτουργίας και να έχει και μεγαλύτερη σημασία η δική μας δουλειά στη δική του όλη αυτή η συζήτηση για τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα ανάλογα με την παρουσία ή την απουσία του Frontex από κάποιες ε, περιοχές και καταστάσεις. Είναι δύσκολο αυτό να εκτιμηθεί. Σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε και περιμένουμε ο Frontex να παίξει ένα ρόλο με συγκεκριμένα πρότυπα και πολύ καλύτερο έλεγχο. Σε άλλε περιπτώσεις αυτό δεν είναι δεδομένο ούτε εγγυημένο ότι θα γίνονται πάντα σεβαστά ή θα πρωταγωνιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χαίρομαι για αυτό που είπατε για τις εκθέσεις ε, της ΥΠΑ της Αρμοστίας και τις επιστροφές και τη φύλαξη των συνόρων. Ε, το είπε όμως και ο Στέφαν, εμείς δεν είμαστε ελεγκτικό όργανο, δεν παρακολουθούμε ε, κάποια ε, λειτουργία κάποιου οργανισμού, ούτε εποπτικό είμαστε. Τελικά ο Frontex ο ίδιος, εμείς συμβουλευτικό όργανο είμαστε. Ο Frontex είναι εκείνος που έχει αυτή την ευθύνη. Εμείς προτάσεις κάνουμε για μηχανισμούς, για μέτρα, έτσι ώστε ας πούμε ο μηχανισμός καταγγελιών που προβάλλεται ως ένα από τα στοιχεία που έχει και τις δυνατότητες ο οργανισμός να αγκιάται τα θεμελιώδη δικαιώματα, κατά πόσο λοιπόν αυτό χρησιμοποιείται με τρόπο σωστό και όσοι ε, βλέπουν τα δικαιώματα τους να παραβιάζονται να έχουν κάπου να προσφεύγουν. Για το θέμα των ανηλίκων επίσης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες οι συστάσεις μας για το ποιο είναι ο ρόλος του καθενό η ευθύνη, η παρακολούθηση, σύστημα αξιολόγησης, ε, κατανομή των ε, πόρων. Ελπίζω φέτος αυτό να γίνει με τη νέα στρατηγική θεμελιωδών δικαιωμάτων και να βρεθεί ένας τρόπος να ε, ασχοληθούν και με τα δικαιώματα των ανηλίκων. Και θα συζητήσουμε με τη Frontex, συνεχίζονται οι συζητήσεις και ε, πάλι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω αν απάντησα, αν τα κάλυψα. Προσπάθησα να καλύψω αυτά που μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν τελειώνει εδώ αυτή η συνεργασία. Α, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι. Ο κύριος Κέσλερ για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι η αρμόδια επάλληλος εκεί και η υπηρεσία ε, το Frontex ε, ότι δεν κάνει δουλειά, ότι δίνεται αυτή η εντύπωση. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Ε, θαυμάσιο το έργο και καταπληκτικό. Αλλά είναι και ενισχυμένη η εντολή τη τώρα και οι δραστηριότητε και η δράση ε, τη υπηρεσία αυτή. Και αγωνίζεται η αρμόδια για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το ευρύ φάσμα το Χρειάζεται και περισσότερο προσωπικό και, και ειδικευμένο προσωπικό για να καλύψει καλύτερα αυτό το ευρύ φάσμα που έχει πλέον. Και δεν δύναται αυτή τη στιγμή να ανταποξέλθει. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε για την παρουσία σας και για την παρουσίασή σας. Απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Και όπως πρότεινε και η Σκά Κέλλερ, θα ζητήσουμε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής μας να απευθύνει επιστολή αρμοδίως και να αναφερθεί και στα θέματα τα πρακτικά των πόρων ανθρωπίνων και οικονομικών. Θα συντάξουμε ένα σχέδιο επιστολής για να το σχολιάσουν και οι συνάδελφοι. Και θα ήθελα να προτείνω κάτι στους συναδέλφους. Είναι γεγονό ότι πολύ συχνά μας αρνούνται την πρόσβαση σε κάποια έγγραφα επικαλούμενοι το απόρριτο ή το εμπιστευτικό για πάρα πολύ καλούς λόγους. Ναι, το ξέρω. Καμιά φορά υπάρχουν και καλοί λόγοι, καμιά φορά είναι πάρα πολύ κακοί λόγοι. Ο κάθε βουλευτής από εμά, όπως και κάθε πολίτης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στην ενημέρωση και αν του την αρνηθούν να προσφύγει σε δικαστήριο. Αν έχετε ειδικά αιτήματα ε, για ειδικέ πληροφορίε, ζητήστε τα και θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε πάνω. Okay, colleagues, that brings us uh, a little later than... Αδελφοί, με μια μικρή καθυστέρηση προχωράμε. Νομίζω θα αναπληρώσουμε τον χρόνο. Περνάμε στα σημεία 4 και 5. Δηλαδή, τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 και μια ανάλογη συμφωνία με την Ελβετική Συνομοσπονδία. Οι δύο εισηγητές απουσιάζουν. Ο κύριος είναι ο Πριμ Ντελβίστησεν του ECR, ο οποίος κολλείεται. Και ο δεύτερο ηγητής είναι ο Κλοντ που επίσης απουσιάζει. Ο κύριος ε, Βίστισεν ε, ζήτησε από το Προεδρείο να διαβαστεί ακόλουθη δήλωση σύμφωνα με τον κανονισμό 515-2014 οι χώρες που σχετίζονται με την εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου Σέγγεν συμμετέχουν ε, στο μέσο χρηματοδοτικής στήριξης ε, συνόρων και θεωρήσεων για να υπάρχει η απαραίτητη δυνατότητα χρηματοδότησης του προπολογισμού του μέσου αυτού στις συνδεδεμένες χώρες και για να καθοριστεί η συνεισφορά της Ισλανδίας στον προπολογισμό. Κατά την άποψη του εισηγητή, έτσι θα επιτευχθεί ένας βασικός στόχος του κεκτημένου Σέγγεν, δηλαδή να μοιραστούμε την ευθύνη για ένα υψηλό αποτελεσματικό επίπεδο ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα για να διασφαλιστεί αφενός η ενιαία στα εξωτερικά σύνορα, με συγχωρείτε, περιλαμβανομένη στις αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και από την άλλη η ομαλή διέλευση των συνόρων σύμφωνα με τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο εισηγητής συνιστά να δώσει το Κοινοβούλιο την συμφωνή γνώμη του το Αυτή ήταν η άποψη του κυρίου Βίστισεν Σε σχέση με την Ελβετία και για την οποία είναι υπεύθυνη ο Βίστισεν. Ε, επίσης ο Κλοντ Μωραές ε, κάνει την ίδια σύσταση. Να συμφωνήσουμε δηλαδή το στόμα και ελπίζω να συμφωνούν και οι σκιώδεις εισηγητές. Θέλει κάποιος τον, τον, τον λόγο, με συγχωρείτε. Κύριε Ντεπχέ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω μόνο να πω ότι συμφωνώ πολύτος και με τους δύο εισηγητάς. Ωραία. Ωραία δήλωση κάνατε. Άλλος? Όχι. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 16 Μαΐου. Μόνο διαδικαστικές τροπολογίες δεχόμαστε στις 12 το μεσημέρι. Η δε ψηφοφορία έχει προβλεφθεί για τις 24 ε, Μαΐου. Α, μήπως θέλει να μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Συμφωνείτε όλοι, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος. Είστε ικανοποιημένοι. Ωραία. Και ερχόμαστε μέσω στο σημείο 6 της μέρης της διάταξης. Αλλά δεν είδα τον κύριο Χρυσόγωνο, ο οποίος είναι εδώ όμως. Ε, σημείο 6. Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών. Ε, proposed... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου του 2017 έκανε μια πρόταση κανονισμού για να απαγορευθούν οι εισαγωγές πολιτιστικών αγαθών που έχουν παρανόμως εξαχθεί από τις χώρες τους που συνδέεται με φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ε, νομιμοποίηση ε, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ΙΜΚΟ και η ΙΝΤΑ είναι επί της ουσίας αρμόδιες. Συγητής μας είναι ο κύριος Χρυσόγονος, τον οποίο η κυρία Σπινέλη όμως απασχολεί. Σταματήστε να απασχολείτε τώρα συντάκτη της νομοδότησής μας, κυρία Σπινέλη. Ο κύριος Χρυσόγονος έχει το λόγο, παρακαλώ. Uh, dear uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πολιτιστικά αγαθά και πολιτιστική κληρονομιά έχουν μια ανεκτήμητη κοινωνική, πολιτική, οικονομική, περιβαλλοντική αξία και είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη μνήμη και την ταυτότητα των πολιτών και δημιουργούν επίσης την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι μία μη ανανεώσιμη πηγή, μοναδική, η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε να υποκατασταθεί, δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με κάτι άλλο και αντιμετωπίζει πάρα πολλές σοβαρές απειλές που έχουν να κάνουν με πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Η παράνομη διακίνωση τέτοιων αγαθών, η αρχαιοκαπηλεία, η λελασία συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, με το ξέπημα βρώμικου χρήματος και με την τρομοκρατία. Προβλέπεται ότι η παράνομη αυτή αγορά αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς αποτιμάται σε 6 με 8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως Επομένως θα λέγαμε ότι είναι η μεγαλύτερη παράνομη αγορά μετά τα ναρκωτικά και μετά τα όπλα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι υπάρχουν αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η ISIS χρησιμοποιούν την παράνομη αυτή αγορά πολιτιστικών αγαθών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Έργα τέχνης και πολιτιστικά αγαθά λοιπόν λαιλατούνται από το ISIS στη Συρία, το Ιράκ, την Ιεμένη και άλλες χώρες οι οποίες πλήττονται από ένοπλες σειράξεις και πολύ συχνά εν συνεχεία τα αγαθά αυτά πολλούνται από οίκους δημοπρασίας στην Ευρώπη, μολονό ότι υφίστανται κανόνες που θα έπρεπε να απαγορεύουν την εισαγωγή αγαθών από τις χώρες αυτές υπό συγκεκριμένε συνθήκες. Μία ιδιαίτερα προβολημένη περίπτωση έχει να κάνει με την πόλη της Παλμύρας, με, τα, ε, με την αρχαιοκαπηλεία πολιτιστικών αγαθών από την πόλη αυτή. Ξέρετε ότι ε, τα πολιτιστικά αυτά αγαθά αποτιμούνται σε πολύ μεγάλα ποσά και υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι αγοραστές, επομένως αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο της παράνομης ε, πώληση τέτοιων αγαθών. Δυστυχώς, λόγω των πολλών διαφορετικών διάβλων πρόθεσης των αγαθών αυτών δεν είναι εύκολη η παρακολούθηση. Η λαιλασία, η αρχαιοκαπηλεία και η παράνομη πώληση των αγαθών αυτών θα πρέπει να ρυθμιστεί περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλέ διαφορετικέ εθνικέ δικαιοδοσίε με πολλού διαφορετικού κανόνε ω προ το δίκαιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται στι ε, διασυνοριακέ ε, δικαστικέ διαφορέ όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά και πολλέ φορέ χρησιμοποιείται και διαφορετικό σύστημα για να καθοριστεί τελικά ένα πολιτιστικό αγαθό αποτελεί όντω αντικείμενο αρχαιοκαπηλεία ή όχι. Αυτή τη στιγμή το εφιστάμενο καθεστώ το οποίο ισχύει για την επιστροφή τέτοιων λιλατηθέντων πολιτιστικών αγαθών είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι ιδιαίτερα κατακαιρματισμένο. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη μας όλους αυτούς τους παράγοντες, συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε το χύτερο δυνατό το ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να καταφέρουμε να επιστρέφουμε τα λιλατιθέντα αυτά πολιτιστικά αγαθά. Αυτή τη στιγμή πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την η εισαγωγή πολιτικών αγαθών θα είναι, βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση, αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό να καλύπτεται επαρκώ η λαιλασία, η αρχαιοκαπηλεία, η παράνομη διακίνηση τέτοιων αγαθών που πολλές φορές καταλήγουν σε βιβλιοθήκες, σε μουσεία ή σε δημόσια αρχεία. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθείτε η προέλευση των αγαθών αυτών. Πολλές φορές έχει να κάνει με ένοπλες διενέξεις, έχει να κάνει με τη δραστηριότητα τρομοκρατικών οργανώσεων. Όλες αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να εντοπίζονται και να τιμωρούνται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να καταπολεμήσουν το παράνομο εμπόριο και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από ένοπλες διενέξεις ιδιαίτερα, από, ιδιαίτερα για τα πολιτιστικά αγαθά εκείνα τα οποία διακινούν τρομοκρατικές οργανώσεις ή άλλες εγκληματικές οργανώσεις. Θα πρέπει να προβλέπεται η επιστροφή των έργων αυτών, θα πρέπει να απαγορεύεται η διαστοριακή διακίνηση τέτοιων πολιτιστικών αγαθών, όπου τα κράτη-μέλη έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι τα αγαθά αυτά προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες και ότι τα έχουν διαχειριστεί, τα έχουν πουλήσει εγκληματικέ ή τρομοκρατικέ οργανώσει και τα οποία δεν υπάρχουν επίσημα πιστοποιητικά. Προκειμένου υπάρχουν ομοιόμορφε συνθήκε για την εφαρμογή του προτινόμενου αυτού κανονισμού, θα πρέπει οι εκτελεστικές αρμοδιότητες να προβλέπονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να προβλέπεται η προσωρινή αποδοχή και αποθήκευση των πολιτιστικών αυτών αγαθών. Θα πρέπει να προβλέπονται ενιαίοι μορφότοποι, ενιαία έγγραφα, καθώς επίσης και ομοιόμορφοι κανόνες για την επεξεργασία των αγαθών αυτών. Θα πρέπει οι εκτελεστικές αρμοδιότητες να έχει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δημιουργηθεί μία αξιόπιστη ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αποθήκευση των αγαθών αυτών και για την ανταλλαγή πληροφοριών για τα αγαθά αυτά μεταξύ των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί διαφάνεια και δημοκρατία, οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να προβλεφθούν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού προηγηθεί διαβούλευση με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να γίνει διαβούλευση και σε επίπεδο γνωμόνων Και αυτή η διαβούλευση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα όριο 250, 250 ετών για τα πολιτιστικά αγαθά, το ελάχιστο αυτό κατόφλι. Εγώ θεωρώ ότι δεν αρκεί το χρονικό αυτό κατόφλι προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία διακινούνται παρανόμως, καθότι θα πρέπει να καταφέρουμε να καλύψουμε όλα τα πολιτιστικά αγαθά, ιστορικά αγαθά, καλλιτεχνικά αγαθά τα οποία δημιουργήθηκαν καθ' όλη την διάρκεια της ιστορίας. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα όριο τουλάχιστον 255 ετών. Προκειμένου να αποφύγουμε το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών, η η απελευθέρωση των αγαθών αυτών και το να περάσουν ουσιαστικά σε ένα καθεστώς ελεύθερης διακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αυτό να γίνεται μόνο μέσω επίσημης δήλωσης στις τελωνικές αρχές της χώρας εισόδου. Σε αντίθεση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ε, ειδικέ ε, σπάνιε συλλογέ, καθώ επίση και είδη χλωρίδα σπανίδας. Θα πρέπει επίση να προβλέπονται πολιτιστικά αγαθά τα οποία έχουν να κάνουν με την φυσική επιστημονική ιστορία, στρατιωτική ιστορία και θα πρέπει να προβλέπονται επίσης νομίσματα, επιγραφές ή άλλα αντικείμενα τα οποία παρουσιάζουν ε, καλλιτεχνικό ιστορικό ενδιαφέρον. Μολονότι μπορεί να αυξηθεί η γραφειοκρατία κατά αυτόν τον τρόπο, θεωρώ ότι η μέθοδος αυτή, η προσέγγιση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να ασφαλίσουμε ασφάλεια και διαφάνεια και να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση και εμπορία πολιτιστικών αγαθών. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει μια δήλωση από τον εξαγωγέα όπου θα εχνηλατείται η όλη διαδρομή των αγαθών αυτών και όπου θα φαίνεται τελικά ότι τα αγαθά αυτά και ότι, ότι, τα αγαθά αυτά πιστοποιούνται ως πολιτιστικά αγαθά σύμφωνα με, τις, με το πλαίσιο της UNESCO. Η προσωρινή αποθήκευση των πολιτιστικών αυτών αγαθών στο, στην τηλεονική επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη στιγμή μπουν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να γίνεται και σύμφωνα με τα ε, λέγονται στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 3 σε περίπτωση κατάσχεσης ή προσωρινής κράτησης πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει να προβλέπονται τα αγένεια για την καλύτερη δυνατή διατήρησή του σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Νοσιακό Δίκαιο. Τώρα, όσον αφορά την κατάλληλη παρακολούθηση και επιτήρηση των ε, αρχαιολογικών πολιτιστικών χώρων, ιδίω ε, για τι χώρε εκείνε που πλήττονται από φυσικέ καταστροφέ ή διενέξει, τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουν περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δοφορική Παρακολούθηση, καθώ επίση και το παρατηρητήριο παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω παράνομη διακίνηση και εμπορία των αγαθών αυτών και προκειμένου να προστατευθεί και η ζωή των πολιτών. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών θα πρέπει επίσης να προβλέπονται κατάλληλες υπηρεσίες, τηλεφωνικές και άλλες, προκειμένου να ενημερώνονται οι αγοραστές πολιτιστικών αγαθών ή άλλοι ενδιαφερόμενοι για το τι συμβαίνει σε σχέση με συγκεκριμένα πολιτιστικά αγαθά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να μην αποκλίνουν από τους κανονισμούς αυτούς και τις ρυθμίσεις αυτές που θα προβλέπει ο προτινόμενος κανονισμός. Ο συντάκτης γνωμοδότησης είμαι στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και να απαντήσω σε ερωτήσεις σας, προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Δύο συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, Κέστερ και Γκόμες. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Χρυσόγονε, σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Η Κομισιόν υπέβαλε μια έκθεση για να καταπολεμήσει την χρηματοδότηση τρομοκρατίας ε, μέσω Τη διακίνηση ε, πολιτισμικών αγαθών. Βεβαίω αυτό είναι ουσιαστικό, αλλά δεν μπορεί να είναι ο μόνο λόγο αυτό η καταπολέμηση τη τρομοκρατία για να σταματήσει αυτό το οργανωμένο έγκλημα. Είναι η κοινή μνήμη του παρελθόντος πολιτισμού που κινδυνεύει από αυτό το εμπόριο. Γνωρίζουμε ότι Υπάρχει μια σημαντική αλλά άγνωστη ποσότητα αρχαιοτήτων στην αγορά που προέκυψε από λάθρα ανασκαφές ε, ή πλιάτσικο σε χώρες ε, που ήταν εμπόλεμες. Αυτό σημαίνει απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα και την πολιτισμική μνήμη γενικώ. Όταν αφαιρούνται από το πλαίσιο οι αρχαιότητες, ο πληθυσμός στερείται τα ήθη και τα έθιμα του. Έτσι καταστρέφεται η πολιτισμική μνήμη μιας περιοχής του κόσμου. Το σπάσιμο αυτού του δεσμού που ενώνει συνεισφέρει στην περαιτέρω αποσύνθεση που προκαλεί ο πόλεμος και ενισχύει τους κρατούντες. Τα λειλατιμένα αντικείμενα επίσης ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιστημονική έρευνα. Η λαιλασία αρχαιολογικών τόπων συνέβαινε παλαιόφεν πριν καταρρεύσει η Συρία, το Ιράκ και η Αίγυπτος, αλλά τώρα πλέον έχει φτάσει σε βιομηχανική κλίμακα. Όσον είναι δυνατόν να γίνεται επικερδές εμπόριο από λάθρανα σκαφές, χωρίς ουσιαστικό κίνδυνο, οι ανασκαφές και οι λελεσίες αυτές θα συνεχιστούν στο μέλλον. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει προστασία ε, εκεί όπου έχουν ζήτηση αυτά τα αγαθά, δηλαδή μεταξύ άλλων στην αγορά των ιδιωτικών συλλογών στην Ευρώπη. Οπότε δεν θα πρέπει να περιστραφούμε μόνο γύρω από τις εισαγωγές, αλλά να δούμε και ποιος θα πρέπει να έχει το θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης σε αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς. Ε, θα πρέπει να είναι το κοινό, κατά την άποψή μου. Οποιαδήποτε συζήτηση για αυτό το θέμα πρέπει να περιλαμβάνει το εάν η ιδιωτική κατοχή αρχαιοτήτων είναι καν αποδεκτή χωρίς ιδιώτες συλλέκτες η μαύρη αυτή αγορά η οποία ασχίζει την συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας θα καταρρεύσει. Χωρίς ιδιωτικές συλλογές τα αντικείμενα αυτά θα τα βλέπει το κοινό μόνο για αισθητικούς λόγους. Ποιος είναι ο άλλος λόγος κατοχής αρχαιοτήτων. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προστατεύσει την πολιτισμική κληρονομιά του κόσμου και θέλει αυτό να επεκταθεί και στις εγκληματικές δραστηριότητες προς όφελος των Ευρωπαίων, τότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αμφισβητήσουμε την ιδιωτική κατοχή πολύτιμων αρχαιοτήτων, έχοντας αυτά κατά νου η λύση που προτείνει η Κομισιόν δεν επαρκεί. Κύριε Κέστερ, να σας ζητήσω... Ε, ναι, ναι, ολοκληρώνω. 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Στις περισσότερες χώρες προέλευσης από τον 10ο αιώνα είναι παράνομη η ιδιωτική κατοχή αρχαιοτήτων. Οπότε δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια δίωδο ελαφρώς νόμιμης κατοχής ε, και ελπίζω η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Θα μπορούσα να προσυπογράψω όλα όσα είπε ο προλαλής σας συνάδελφος Κέσνερ, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο μας χρειάζεται ε, να αναλάβουμε δράση κατά ε, του λαθρεμπορίου αρχαιοτήτων. Υπάρχει όμως, είναι σημαντικός αυτός ο λόγος κατά πολέμης τρομοκρατίας, γιατί γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας έχει βρει ένα τρόπο τώρα να εκμεταλλεύεται την αρχαιοκαπηλεία και σε χώρες όπως είναι η Συρία, το Ιράκ και πρόσφατα η Λιβύη, όπου λαιλατούν αρχαιολογικούς χώρους για να χρηματοδοτούν την τρομοκρατική τους δραστηριότητα. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι λόγοι, τους οποίους αναφέρατε κι εσείς, που συνεγορούν υπέρ της δικής μας ενασχόλησης. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον ε, συντάκτη της νομοδότησής μας, να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε Θέλω να τον ευχαριστήσω για την ε, γνωμοδότηση αυτή και να τον ρωτήσω το εξής. Έχετε σκεφτεί και το ρόλο των ελευθέρων λιμένων. Των ελευθερών ζωνών. Όπου αποθ... έτσι, να αποθηκεύονται στα λιμάνια αυτά τα αγαθά μέχρι να διευκρινιστεί η προέλευσή τους και το εμπόριο στα πλαίσια της Επιτροπής ε, για τα έγγραφα του Παναμά έχουμε αρχίσει να το εξετάζουμε αυτό. Πήγαμε και στο Λουξεμβούργο για να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ελεύθερες ζώνες και τις ατέλειες. Και ποιος υποτίθεται ότι τα ελέγχει όλα αυτά στο Freeport Luxembourg. Και περιμένουμε τις απαντήσεις που δεν λάβαμε ακόμα. Και στη Γενέβη υπάρχει μια τεράστια ε, ζώνη ε, ε, φορολόγητη. Είναι παντού το θέμα αυτό, διάχυτο και χρειάζεται οπωσδήποτε να ασχοληθούμε. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις ελεύθερες ζώνες όπου φυλάσσονται, αποθηκεύονται από τους ιδιοκτήτες, τους διακινητές τους τα αγαθά αυτά και φεύγουν κάθε ελέγχου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή θα πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση και της δημοκρατίας και των παρανόμων δραστηριοτήτων. Κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξή. Να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε όταν εντοπίζονται αυτές οι αρχαιότητες στην Ευρώπη. Κυκλοφορούν ήδη λαθρέα αρχαία. Τις βρίσκουν λοιπόν οι κρατικές αρχές, αλλά δεν μπορούν να επιστρέψουν τα αρχαία αυτά στις πατρίδες τους γιατί δεν έχει κυβέρνηση ας πούμε η Λιβύη. Πρόσφατα ξέρουμε ότι υπήρξε ένα δίκτυο που αποκάλυψε η ε, Ισπανική αστυνομία όπου διαλεύκανε ένα τέτοιο λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων από τη Λιβύη. Λοιπόν, αυτό αποκαλύπτεται. Κάποια κρατική αρχή δεν θα πρέπει να τα προστατεύσει αυτά, γιατί είναι κληρονομιά της ανθρωπότητας, μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν σε μια χώρα που θα μπορεί να τα προστατεύει σωστά, γιατί θα έχει σωστή διοίκηση, πράγμα που δεν συμβαίνει δυστυχώς ακόμα αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Ευχαριστώ πολύ. Πριν επανέλθουμε στον κύριο Χρυσόγωνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσθέσει τίποτα στην παρούσα φάση. Έχετε. Σύντομα σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ γρήγορα μερικά πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ για τις τροπολογίες. Θα τις λάβουμε υπόψη μας. Αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να βελτιώσουμε την πρόταση. Πολύ λίγα πράγματα για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Το άρθρο 207 της συνθήκης που είναι η παρούσα νομική βάση δεν το καλύπτει αυτό. Και δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο νομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να νομοθετήσει για την επιστροφή από ένα κράτος μέλος σε τρίτη χώρα ενός ε, κατασκευέντος αντικειμένου. Υπάρχει σύμβαση της UNESCO που διέπει ε, αυτή την επιστροφή και μέχρι σήμερα αυτό γίνεται δια των διπλωματικών οδών. Έτσι επιστρέφουν στις χώρες τους. Um, we, Λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι προτείνει ο εισηγητής τα 75 έτη ως ελάχιστη ηλικία το τόριο. Εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα για επιπλέον κατηγορίες που προσθέσατε, που προτείνατε να βγει ε, ε, ε, υποχρέωση άδειας εισαγωγής, ιδιαίτερα η κατηγορία Α, ε, παλαιοντολογικά είδη ή χλωρίδα και πανίδα δεν είναι ακριβώς πολιτιστικά αγαθά γιατί δεν είναι κάτι το οποίο έχει ε, δημιουργήσει ο άνθρωπος και τα παλαιοντολογικά αγαθά ε, καταλαβαίνετε και λόγω ηλικία τι συμβαίνει εκεί. Θα τα εξετάσουμε όλα αυτά. Very much. Uh, Υποστηρίζουμε πάρα πολύ ότι είπαν οι ομιλητές Όλα αυτά τα γράφει και το μνημόνιο. Μάλλον η αιτιολογική έκθεση και η μελέτη που έχουμε εκπονήσει για τον αντίκτυπο της πρότασης. Το έχουμε σκεφτεί αυτό το θέμα των ελευθέρων ζωνών, των αφορολογήτων ε, Προβλέπεται αυτό στο κείμενο και για τις άδειε. και για τέτοιε τέτοιες ελεύθερες περιοχές που δεν έχουν ε, δασμούς, ε, φορολογική ή δασμολογική ατέλεια. Στο άρθρο 3 νομίζω αναφέρεται μια τέτοια διάταξη ε, για έκτακτες ανάγκες όπου δεν μπορούν να επιστρέψουν τα αγαθά αυτά κάπου να αποθηκεύονται προσωρινά από μια κρατική αρχή μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση και η ομαλότητα σε μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη σύραξη ας πούμε. Ευχαριστώ. Ε, σε επανέλθουμε λοιπόν στον ε, συντάκτη της νομοδότησης. Σύντομα παρακαλώ κάποια καταληκτικά σχόλια. εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν την συζήτηση για τις πολύ οικοδομητικές παρατηρήσεις και να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τροπολογίες είναι 22 Μαΐου στις 12 η ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Έτσι περνάμε στα σημεία 7 και 8 τα οποία έχουν αναβληθεί, οπότε δεν θα τα συζητήσουμε σήμερα, αλλά περνάμε στο σημείο 9, που είναι δικό μου αίτημα. Δηλαδή το θέμα της ε, γραπτής ερώτησης που υπέβαλα στις ε, κομισιόν, στην Κομισιόν με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου για τον Ιταλικό νόμο περί εξαετούς υποχρεωτικής διατήρησης δεδομένων των τηλεπικοινωνιών για ένα ελάχιστο διάστημα 6 ετών. Και ενδιαφέρον είναι ότι αυτό εγκρίθηκε στο πλαίσιο ενός νόμου στροπολογία, δηλαδή σε έναν νόμο περί ηλεκτρικών σκουπών. Λίγο περίεργος τρόπος νομοθεσίας. Εν τω μεταξύ η Κομισιόν απάντησε, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να ενημερωθεί και η Επιτροπή για να μας απαντήσει η Κομισιόν. Γιατί η Κομισιόν είπε βεβαίως αυτά είναι εθνικές υποθέσεις, δεν είναι δική μας δουλειά. Και νομίζω ότι η Κομισιόν προετοιμάζει μια νέα νομοθετική πρόταση για μια νέα οδηγία διατήρησης ε, των δεδομένων. Έξι χρόνια εμένα μου φαίνονται πάντως υπερβολικά και αντίθετα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θέλω να ακούσω λοιπόν την Κομισιόν. Νομίζω ότι έχουμε την κυρία Φακλέη η οποία είναι βοηθός ε, τμήματάρχης του αρμόδιου τμήματος. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για την πληρότητα όμως της υπόθεσης θα επαναλάβω την απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος ο κύριος Αβραμόπουλος. Στο πρώτο τμήμα της ερώτησής σας η Κομισιόν απάντησε ότι γνωρίζει τον Ιταλικό νόμο και θα λάβει την απόφαση κατόπιν της αναγκαίας αναλύσεως την απόφαση για το αν θα ξεκινήσει μια διαδικασία παραβάση. Για το δεύτερο μέρος της ερώτησής σας, Κομισιόν απάντησε πως η εποπτεία αυτής της νομοθεσίας είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, συγκεκριμένα των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαστηρίων. Για το τρίτο και τελευταίο τμήμα της ερώτησής σας η απάντηση ήταν ότι ε, δουλειά στο θέμα αυτό συνεχίζεται κατόπιν ε, της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην περίπτωση ΤΕΛΕ 2. Στην απόφαση στην οποία συμμετέχει και η Κομισιόν ε, μαζί με τα κράτη-μέλη και τέλος, όπως είχε πει και στο πρόγραμμα εργασίας του 2018, η Κομισιόν θα ολοκληρώσει το τι θα κάνει όσον αφορά τις κατευθύνσεις που θα δοθούν στο ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Έχω ήδη δύο αιτήματα, αλλά ως συντάκτης ε, της ερώτησης, ε, να σας κάνω μια ερώτηση επιπλέον για να απαντήσετε. Λέτε ότι επαφίεται στις εθνικές αρχές. Το θέμα είναι ότι έγιναν αυτές οι συστάσεις ε, προς ε, την χώρα για να μην εφαρμοστεί ο νόμος αυτός. Οπότε αυτό το οποίο μπορεί να κάνουν οι πολίτες είναι μόνο να προσφύγουν στα δικαστήρια, κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Και βεβαίως ε, δεν είναι αυτός κατάλληλος τρόπος προστασίας ε, των δεδομένων δηλαδή ο θεματοφύλακας των συνθήκων να λέει να πάνε οι πολίτες στα δικαστήρια. Θα σας αφήσω να το σκεφτείτε, εν πάση περιπτώσει, και εν τω μεταξύ έχουν ζητήσει τον λόγο η κυρία Σπινέλη και Ζίπελ. Κυρία Πρόεδρε, Σοφή, θα ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω για την ερώτηση αυτήν που υπέβαλες, ερώτηση η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί έχει να κάνει και γενικότερα με το κράτος δικαίου και την ένωμη τάξη στην Ιταλία. Η απάντηση του Επιτρόπου Αβραμόπουλου πραγματικά δεν με ικανοποιεί καθόλου. Νομίζω ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές αρμοδιότητες εδώ συνδέονται άμεσα, γιατί μιλάμε άλλωστε για ευρωπαϊκούς νόμους εδώ. γιατί βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει η Ιταλική νομοθεσία που αυξάνει σε έξι έτη την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων. Ο Αντωνέλο Σόρο, που είναι ο υπεύθυνο τη Αρχή Προστασία Δεδομένων στην Ιταλία, αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή την νομοθετική και νομίζω ότι αντιβαίνει ούτως ή άλλως την ομολογία και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίω στην υπόθεση Τελεντούε του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούν να, αποδεχθούν, να γίνουν αποδεκτές εθνικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν είναι αναλογικές και οι οποίες δεν είναι περιορισμένες στο χρόνο. Και καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σοβαρό για την Ιταλία, γιατί ουσιαστικά στο όνομα της έκτακτης κατάστασης που μπορεί να έχει να κάνει με την καταπολέμηση της μαφίας ή της τρομοκρατίας, κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή να επισημοποιήσουμε και να μονιμοποιήσουμε νόμους που θα έπρεπε να έχουν καθαρά προσωρινό χαρακτήρα. Και ο ίδιος ο επόπτης της προστασίας δεδομένων στην Ιταλία παρέπεμψε στην απόφαση Τελεντούε του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται οι δυσανάλογες περίοδοι διατήρησης δεδομένων. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν θεωρώ ότι ε, πρέπει πραγματικά εδώ πέρα να γίνει κάτι. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα διαδικασία επί παραβάση, όπως προτείνει άλλωστε η ερώτησή σου. Θεωρώ ότι πραγματικά τίθεται να αμφιβόλω εδώ πέρα η ίδια η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει λόγος να επικρίνουμε άλλες χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και να διστάζουμε αυτή τη στιγμή να λάβουμε δράση κατά της Ιταλίας που παραβιάζει τελικά το νοσιακό δίκαιο μέσω των αποφάσεων της αυτών. Κυρία Σίπελ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και θα πρέπει να φύγω αμέσως μετά την παρέμβασή μου αυτή, γιατί έχω μια άλλη συνάντηση εκτός Κοινοβουλίου. Θεωρώ πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Η Ιταλική αυτή νομοθεσία έχει ένα ολόκληρο ιστορικό, θα έλεγα και η υποχρεωτική αυτή διατήρηση δεδομένων που προβλέπεται είχε απασχολήσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο παρελθόν. Έχουμε τώρα τη νέα αυτή διαδικασία, την αφέρατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, μια νέα διαδικασία που δίνει την εντύπωση πραγματικά ότι η Ιταλική κυβέρνηση δεν ήθελε να ανοίξει εκ νέου το ζήτημα της διατήρησης των δεδομένων, κατάφερε να κρύψει πάρα πολύ καλά τη νέα αυτή νομοθετική διάταξη ω τροπολογία σε έναν άσχετο νόμο, όπως είπατε κι εσείς. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε καταρχάς την βάση του νόμου αυτού, άρθρο 20 για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική νομική βάση αυτής της νομοθεσίας. Ακόμα και στο προήμιο της σχετικής αυτής κοινοτικής οδηγίας για την καταπολέμηση τρομοκρατίας, δηλαδή μιλάμε για την ε, αναλογικότητα. Και μιλάμε επίσης και για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχουμε λοιπόν πολλούς λόγους ε, για να απορρίψουμε τελικά την τελική αυτή με το βασικό επιχείρημα ότι δεν συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία, δεν συνάδει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Δεν μπορώ λοιπόν πραγματικά να καταλάβω για ποιο λόγο η μόνη απάντηση που μας δίνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Μα αν το πω αυτό εγώ στους πολίτες, στη δική μου εκλογική περιφέρεια θα μου πούνε ναι. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινέ αξίε και κοινού κανόνε. Πώς μπορούμε λοιπόν ξαφνικά να μιλάμε για το ζήτημα αυτό μόνο για εθνική αρμοδιότητα. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει περαιτέρω δράση και να μην κρύβεται πίσω από την απάντηση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πριν φύγετε και δώσω το λόγο στην κυρία Fairplay, θα πρότεινα στους συντονίστες να σκεφτούν μήπως χρειαστεί να ζητήσουν και τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για το επιχείρημα που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει υποτίθεται την εξουσία ή την αρμοδιότητα, την ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Εγώ θέλω κανονική ανάλυση ε, αυτού του επιχειρήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν οφείλει να δώσει συνέχεια και να δράσει. Και ως συντονίστρια ε, σας το θέτω υπόψη και σας το εμπιστεύομαι. Ευχαριστώ κύριε Φερκλέ. Σας ευχαριστώ και πάλι πρόεδρε. Κατανοώ τις ερωτήσεις σας και των άλλων δύο μελών του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα δεν έχει προσφύγει επί παραβάση κατά της Ιταλίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τι περιμένει για να το κάνει. Κοιτάξτε, θα πρέπει να καταλάβουμε και να τονίσουμε ότι οι συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο διατηρούν τα δεδομένα των ε, τηλεπικοινωνιών τα κράτη είναι περίπλοκο θέμα και μετά από την αντίστοιχη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι ευρύτερη συζήτηση και είναι πάγια τακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση για προσφυγή επί παραβάση που είναι βαριά και σημαντική η απόφαση να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πλήρες επιπτώσεις ε, ε, ε, στα κράτη-μέλη ε, μια τέτοια δικαστικής απόφασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε. Είναι μια πάγια τακτική μας και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη αντικτύπου που κάνουμε με τα κράτη-μέλη, με τη Europol, με το ε, Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με όλους τους αρμόδιους φορείς. Εξετάζουμε τις επιχειρησιακές ικανότητες των διοκτικών αρχών, τα δεδομένα για την προστασία της προσωπικής ζωής και τα λοιπά και το θέμα είναι πιο περίπλοκο από ό,τι περιμέναμε. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει ε, ακόμα προβεί στη συγκεκριμένη απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να κινήσει όχι ε, προσφυγή. Μάλιστα. Θα με αυτή η ανάλυση, γιατί εγώ δεν το βρίσκω τόσο περίπλοκο. Δηλαδή εμένα μου φαίνεται, μα και εσείς στην απάντησή σας μιλάτε για τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια εθνική αρχή λέει ο νόμος αυτός παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ε, πόσο δύσκολο είναι. Κάπου δηλαδή έχω βαρεθεί να ακούω την Κομισιόν. Η μόνη απάντηση που λαμβάνουμε είναι η ίδια. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Όλη παρακολούθηση. <laughs> Εάν οι εθνικές αρχές θεωρούν ότι παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν έχει αρμοδιότητα να δράσει, πρέπει να δράσετε εσείς δηλαδή. Πόσο δύσκολο είναι. Τέλος πάντων. Είναι και πολύ λίγη στην αίθουσα για να γίνει μια πραγματική συζήτηση. Απλά θα ήθελα η Επιτροπή μας να ζητήσει επισήμως μια νομική ανάλυση της κατάστασης και συγκεκριμένα την υποχρέωση της Κομισιόν να επιβάλλει το ευρωπαϊκό δίκαιο. όχι μόνο τη στιγμή που είναι πολιτικά βολικό, αλλά τη στιγμή που παραβιάζεται ο νόμος. Και το συντομότερο δυνατόν αυτή είναι η υποχρέωση της Κομισιόν. Απέναντι στους πολίτες. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. τώρα έχουμε ένα πρόβλημα όμως, γιατί το επόμενο θέμα, το 10, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ε, είναι του κυρίου Κορά, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα. Έρχεται σε δύο-τρία λεπτάκια. Εντάξει, θα αντέξουμε. Wash your hands or get coffee. Πηγαίνετε λίγο στην τουαλέτα, πιείτε κανένα καφεδάκι. Who Ποιος θέλει να μας τραγουδήσει κάτι. We're here so we can start, is that it? Yeah. we're still, apparently the rapporteur is in an elevator somewhere, so he can't be far. Έρχεται ο εισηγητής από ό,τι φαίνεται είναι σε ένα σανσέρ. Φτάνει σύντομα. Of course we can quickly take all sorts of official decisions here now. Στον διάμεσο διάστημα να πάρουμε πολλές επίσημες αποφάσεις. It on the agenda, point Στο σημείο 10 είμαστε, καταφτάνει και ο εισηγητής από ό,τι μου λένε σε ένα σανσέρ. Καταπληκτικά έφτασε και ο εισηγητής. Okay. As taking seat, I will do the introduction. Κάθεται, ας πω κάποια εισαγωγικά λόγια. Ενημέρωση όσον αφορά τις επραγματεύσεις στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου για την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. Ο τέταρτο τριμερή διάλογο έλαβε χώρα στι 12 Απριλίου, επόμενο προβλέπεται για τι 30 Μαου στο Στρασβούργο. Ο κύριο Κορά θα μα ενημερώσει. Σα ακούμε. Πολύ ωραία. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ζητώ συγγνώμη που έφτασα με καθυστέρηση. Είχα καθυστέρηση και με την πτήση μου και έφτασα από την άλλη πλευρά της Ευρώπης. Ε. Λοιπόν, Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου, του κοιόδη συγητές για την προσήλυση και τη δέσμευση που δείξανε κατά τη διάρκεια τη όλη διαδικασία για το σημαντικότατο αυτό νομοθέτημα. Να ευχαριστήσω και την Βουλγαρική Προεδρία για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και τι προσπάθειε που κατέβαλε προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό κοινό αποδεκτό από όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομητική τη στάση που έδειξε και συνεχίζει και δείχνει στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Η βασική αρχή ήταν να καταλήξουμε σε ένα αποτελεσματικό νομοθετικό κείμενο, πλήρες και σαφές, που να κλείσει πραγματικά τα νομικά αυτά κενά τα οποία χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, προκειμένου να προχωρούν σε νομοποίηση εισόδων από εγκληματικέ δραστηριότητες και για να χρηματοδοτούν κατά αυτόν τον τρόπο τις δραστηριότητές τους. Ξέρετε ότι όπως είπε και ο δικαστής Φαλκόνε, τον οποίο δολοφόνησε η μαφία, θα πρέπει πάντα να παρακολουθούμε, να ακολουθούμε τα χρήματα, γιατί εκεί πέρα που βρίσκονται τα χρήματα βρίσκονται και εγκληματίε. Θεωρώ λοιπόν ότι με, την, ε, με το νέο αυτό νομοθέτημα το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταφέρουμε να πετύχουμε ακριβώς αυτό, να παρακολουθήσουμε καλύτερα την ε, οδό που ακολουθούν τα χρήματα και να καταφέρουμε τελικά να καταπολεμήσουμε την ε, νομοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Είχαμε συνεδριάσει σε τεχνικό επίπεδο, έχουμε κάνει τέσσερι τριμερεί διαλόγου και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε στον επόμενο πολιτικό τριμερή διάλογο που θα γίνει στι 30 Μαου στο Στρασβούργο να ολοκληρώσουμε την όλη διαδικασία. Σε λίγε μέρε δηλαδή. Στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου καταλήξαμε συμφωνία για κάποια σημαντικά ζητήματα τις οδηγίες αυτής που θα πρέπει να εφαρμόζεται για όλες τις κατηγορίες εγκληματικών δραστηριοτήτων χωρίς να προβλέπονται παρεκκλήσεις. Προβλέπονται επίσης κοινέ κυρώσεις για τα φυσικά πρόσωπα και προβλέπεται επίσης η απαγόρευση συμμετοχής των νομικών προσώπων σε δημόσιες συμβάσεις. Προβλέπεται επίσης το να υπόψη και επιβαρυντικές περιστάσεις. Επίσης, Σύμφωνα με, με τους ορισμούς που έχουμε στα πλαίσια της οδηγίας θα προβλέπονται πλέον ε, κοινέ προϋποθέσεις προκειμένου να καταλήξουμε σε επιβαρυντικές ε, περιστάσεις ιδίω ε, όσον αφορά την εμπλοκή συγκεκριμένων φυσικών προσώπων σε εγκληματικέ δραστηριότητε και σε νομοποίηση εγκληματικών εσόδων. Ελπίζω ότι τα ζητήματα τα οποία παραμένουν θα επιληθούν πολύ γρήγορα προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να δώσουμε ένα νέο μέσο στις διοκτικές αρχές προκειμένου να είναι σε θέση να τιμωρούν το ιδεχθές αυτό έγκλημα της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτά είχα να σας πω. Σε αυτές τις σημαστικές λύσεις έχουμε καταλήξει μέχρι στιγμής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να πάρει κάποιος άλλος το λόγο. Ο κύριος Σετχόφσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω πολλές ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Ποια είναι τα συγκεκριμένα συμπεράσματα τώρα στα οποία καταλήγουμε. Η έκθεση συγκεκριμένα, τι θα πρέπει να πραγματεύεται και ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε συμβιβασμούς στις διαπραγματεύσεις. Άκουσα ότι κάποια κράτη-μέλη είχαν προβλήματα με την έκθεση. Ξεπεράστηκαν αυτά, τα λύσαμε. Και τελευταία ερώτηση. Ασχοληθήκατε και με το θέμα των εμβασμάτων πολύ μικρών ποσών στα κράτη-μέλη. Συνήθως μαθαίνουμε για τα διασυνοριακά εμβάσματα μεγάλων ποσών. Ασχοληθήκατε με τα μικροεμβάσματα γιατί πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις διακινούν ποσά μικρά, πολύ μικρότερα, τα οποία στέλνουν από λογαριασμό σε λογαριασμό για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε. Άλλος κανείς, όχι. Ο Κοράου. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την ερώτηση αυτή. Δεν είχα βάλει κατευθείαν τα ακουστικά, δεν άκουσα την αρχή της διερμηνίας. Ελπίζω να μην έχασα κάτι από την παρέμβασή του. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι αναφερόμαστε εδώ πέρα σε μία οδηγία που έχει να κάνει με το ποινικό δίκαιο. Δεν μιλάμε λοιπόν γενικά και αόριστα για νομοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Μιλάμε για εναρμόνιση του ποινικού δικαίου των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Και ο στόχο εδώ πέρα είναι οι διοκτικές ρυθμίσεις όσον αφορά την εργασία των διοκτικών αρχών και οι διατάξεις του ποινικού δικαίου να καταφέρουν κάπως να δραμονιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια επίσης οδηγίας αυτής λέμε ότι τα κύρια, κύρια δικήματα, θέλετε, από τα οποία προέρχονται οι νομοποιούμενες πρόσοδοι, θα πρέπει να είναι τα ίδια παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μιλάμε παντού για τα ίδια κύρια αδικήματα, προκειμένου και οι δικαστές να μπορούν να ακολουθούν κοινέ διαδικασίες, να επιβάλλουν κοινέ κυρώσεις. Θέλουμε επίσης να εναρμονίσουμε την ίδια την έννοια του εγκλήματος αυτού, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα και θέλουμε επίσης να καταφέρουμε να επιλύσουμε αυτή τη στιγμή τις διαφορές που μπορεί να προκύπτουν όσον αφορά την δικαιοδοσία, για το ποιο δικαστήριο δηλαδή ποια χώρα είναι αρμόδιο. Και θέλουμε να επιλύσουμε την περίπτωση εκείνη όπου κανένα κράτος μέλος δεν προτίθεται τελικά να εκδικάσει ένα συγκεκριμένο αδίκημα. Και επίση τίθεται και κάποια ευαίσθητα ζητήματα, όπω το ζήτημα τη ε, κατάσχεσης και της δίμευσης. Θέλουμε πάλι εδώ πέρα μία προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματικά να βοηθά τα κράτη-μέλη. Στο ενδιάμεσο διάστημα, περιμένοντας δηλαδή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσσωρευμένη πείρα που έχουν τα κράτη-μέλη για να καταφέρουν να έχουν και στο ζήτημα αυτό της δίμευσης μια κοινή προσέγγιση. Νομίζω ότι επ' αυτού μάλλον θα έχουμε απλώς μία αναφορά στο κείμενο, αλλά ενδεχομένω να μην υπάρχει τελικά μία ενοποιημένη ρύθμιση. Αυτό ενδεχομένω να το κάνει η επόμενη κοινοβουλευτική θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, στα πλαίσια του ποινικού δικαίου θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις διατάξεις εκείνες οι οποίες σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζονται. Πάντως, ως προς τις αρχικές προτεραιότητες που είχαμε θέσει, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι μεγάλη πλειοψηφία στο Συμβούλιο και βέβαια μεγάλη πλειοψηφία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνηση συγκεκριμένων σημείων και κατά αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να ξεπεράσουμε κάποια πρώτα προβληματικά σημεία. Δεν μιλάμε για συγκεκριμένα ποσά αυτή τη στιγμή, γιατί αναφερόμαστε, όπω σα είπα, σε ποινικό δίκαιο, αναφερόμαστε σε κατασταλτικέ δράσει, αναφερόμαστε σε κυρώσει στην όλη διαδικασία που ακολουθείται, δηλαδή στο ποινικό δίκαιο. Γι' αυτό το λόγο δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε συγκεκριμένα ποσά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει να πει κάτι. Όχι. Ωραία. Τελειώνουμε και με αυτό το θέμα. Και φτάνουμε στο σημείο 11, το οποίο θα συζητηθεί και κλεισμένο των θυρών. Οπότε, παρακαλώ, οι μη έχοντες εργασία